ήθελα καταρχήν να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, τον κύριο Νικόλα Σμιτ. Παρακαλώ κύριε Σμιτ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιότιμοι βουλευτές. Μόλις ακούσαμε τον πρόεδρο Γιούνκερ, και όλοι ξέρουμε πως η κατάσταση που ήδη ήταν πάρα πολύ δύσκολη πριν τις καλοκαιρινές διακοπές έχει προσλάβει πλέον καταστροφικές διαστάσεις ε, με αριθμούς ρεκόρ για στις τρεις βασικές οδούς ε, κεντρική και ανατολική Μεσόγειος και δυτικά Βαλκάνια. Διαφοροποιείται δε η τωρινή κατάσταση από τις παρελθούσες ε, λόγω του εύρους της ε, με κλιμακωτές ε, αντιδράσεις επιτόπου και μια σύγχυση άνευ που έχει δημιουργηθεί λόγω αυτών. Η πίεση που ασκείται στις ικανότητες υποδοχής που έχουμε, γλωσσικές και διοικητικές ικανότητες είναι εξαιρετικά υψηλή. Και πέρα όμως από τους αριθμούς ε, και τα θεσμικά ζητήματα, είναι στοιχειώδου σημασία να θυμόμαστε στα πλαίσια αυτής της συζήτησης ότι η κατάσταση πάνω απ' όλα δείχνει ε, ανθρώπινα δράματα, ε, προσωπικές τραγωδίες που εκτιλήσονται και που πλήττουν οικογένειες ολόκληρες. Με την περιπλοκότητα αυτών των ζητημάτων απλή απάντηση δεν υπάρχει και χρειαζόμαστε μια αποφασιστική και συνεκτική απάντηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συνδυάζει αφενός την ευθύνη, αφετέρου την αλληλεγγύη. Οφείλουμε να εφαρμόσουμε μια βιώσιμη κοινή πολιτική για τα μεταναστευτικά ζητήματα. Θα πρέπει να σπεύσουμε προετοιμάζοντας ταυτόχρονα μακροχρόνιες λύσεις, σφαιρικές βιώσιμες λύσεις δοθήσεις της εξωτερικής διάστασης ε, του προβλήματος με το οποίο έχουμε έρθει αντιμέτωποι και ε, δεδομένου του αντικτύπου του ε, στην Ευρώπη, στις σχέσεις που έχουν τα κράτη-μέλη ανάμεσά τους, θα πρέπει να παραδεχτούμε το προφανές ότι δεν πρόκειται να είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε το πρόβλημα εάν δεν συσπηρωθούμε. Επαναλαμβάνω και πάλι αυτά που σας είπα στην προηγούμενη συζήτηση. Η βασική μας μέρημνα θα σχετίζεται με την ασφάλεια των ίδιων των ατόμων. Είναι μια ηθική υποχρέωση που έχουμε, την οποία φέρουμε και δυνάμει του διεθνούς δικαίου. Ε, το ίδιο ισχύει και για όλους τους κρατικούς εφορείς ε, που ε, είναι ε, παρόντες σε, αυτά, σε αυτές τις περιοχές ε, όπου υπάρχουν ένοπλες σειράξεις ή στις χώρες διέλευσης επίσης. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια αξιοπρεπή υποδοχή για όλους όσους θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το καθεστώς παροχής διεθνούς προστασίας. Θα ήθελα να υπενθυμίσω επίσης αυτό που ανέφερε εξάλλου και ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για, αυτές ε, τις αυτά, για αυτά τα δεκάδες εκατομμύρια ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έδειξαν μια καταπληκτική αλληλεγγύη που είναι και η απόδειξη της ικανότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιδείξει ε, αλληλεγγύη και θα ήθελα, όπως είπε και ο ε, Γερμανός Πρόεδρος, ε, να μιλήσω για μια για μια φωτεινή Ευρώπη ε, νομίζω ότι ε, αυτή την Ευρώπη θέλουμε να υποστηρίξουμε, αυτή την Ευρώπη θέλουμε να ε, προωθήσουμε, να σε επιτρέψουμε να προχωρήσει. Για τι ικανότητε υποδοχή θα πρέπει να αναβαθμιστούν τόσο στην να στο ύψο των προκλήσεων τόσο στην επικράτηση Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στι τρίτε χώρε. Χρειαζόμαστε ένα κοινό μέτωπο και καταλαβαίνουμε και τον δημοσιονομικό αντίκτυπο που θα έχουν αυτά τα μέτρα και φυσικά αυτό σα αφορά πρωτίστω στην, στην οδό των δυτικών Βαλκανίων ε, είναι επιλέξιμος επιτοπλίστων οι πρόσφυγες για την παροχή διεθνούς προστασίας. Τους περασμένου μήνε, επανειλημμένα οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων σε αυτό το πρόβλημα, το περίπλοκο ζήτημα ε, των προσφύγων και των μεταναστών και απίφθηναν έκκληση για μια σφαιρική προσέγγιση επικεντρώνοντας την προσοχή τους σε τρεις βασικές διαστάσεις που πρέπει εκ παραλίλου να υποστηριχθούν η ε, μετεγκατάσταση και επανεγκατάσταση, η επιστροφή, επανεισδοχή και επανένταξη, καθώς και η συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης. Σε αυτό τον μήνα Ιούλιο το Συμβούλιο στον τομέα της ε, ε, μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης σημείωσε πρόοδο. Και επειδή μιλάμε τώρα για τα εργαλεία επίγουσας δράσης, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι σήμερα εγκρίνει ε, την έκθεση Keller και χάρη στην οποία την επόμενη Δευτέρα μπορούμε να λάβουμε τις αποφάσεις μετεγκατάστασης και κυρίως, αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία, επανεγκατάστασης όλων όσων έχουν φτάσει από τις 15 Ιουνίου Αυγούστου και μετά. Είναι απαραίτητο αυτό να γίνει για να δώσουμε μία απάντηση στις ανθρώπινες τραγωδίες, στην ανθρωπιστική κρίση που ε, βιώνει σήμερα η Ευρώπη. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις νέες προτάσεις που έχει καταθέσει και που λαμβάνουν υπόψη τα τελευταία γεγονότα και το εύρος κυρίως του προβλήματος. Για τις επόμενες εβδομάδες και επόμενους μήνες η Προεδρία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να σημειωθεί πρόοδος για το σύνολο των προτάσεων και γι' αυτό η Προεδρία μας συνεκάλεσε ένα Συμβούλιο Τζάι έκτατο ε, στις 14 Σεπτεμβρίου την επόμενη Δευτέρα που θα αναθεωρήσει ε, το όλο το φάσμα των μέτρων που πρέπει να αναλυφθούν. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες όμως υπάρχουν άμεσες προτεραιότητες. Η ε, εγκατάσταση των hotspots, η ενίσχυση των αποτελ... της αποτελεσματικότητας των πολιτικών μας ε, για την επιστροφή και για την επανεισδοχή και η καταπολέμηση ε, της δράσης ε, των διακινητών. Για, στο διεθνέ επίπεδο θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μα με του εταίρου μα για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, κυρίω με την Αφρική και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώ βέβαια και με την Τουρκία. Σε αυτή την προσπάθεια Κάθε κράτος μέρος ξεχωριστά και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμβάλλουν μέσα σε ένα πνεύμα υπευθυνότητας και κοινή δράση. Χρειαζόμαστε μια λύση η οποία θα αγγίζει όλα τα ζητήματα, όλα τα προβλήματα. Μία λύση που πραγματικά θα δίνει απάντηση στις προκλήσεις με τις οποίες καλούμεθα πλέον, ε, ε, ε, στις οποίες καλούμεθα να αντεπεξέλθουμε. Έχουμε διαφορετικές παραδόσεις, διαφορετικές εθνικές παραδόσεις. Όμως σήμερα έχουμε το ηθικό καθήκον να κάνουμε την απαιτούμενη υπέρβαση και να επικεντρωθούμε στα κοινά μας στοιχεία, στον κοινό μας παρονομαστή που επικρατεί σε σχέση με τις διαφορές που μας χωρίζουν. Σε αυτό το πλαίσιο υπολογίζουμε στην ενεργό συμβολή και συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με χαρά θα ακούσω τώρα τη συζήτηση που θα ακολουθήσει ε, και σίγουρα θα ε, μεταφέρω ε, τη, τα αποτέλεσμα της συζήτησης στο Συμβούλιο. Όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Σμιτ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον αντιπρόεδρο κύριο Τίμερμαντς. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να μιλήσω διαμακρόν διότι ο πρόεδρος κύριος Γιούγκερ σας εξήγησε διεξοδικά τις προτάσεις και τα προγράμματα της Επιτροπής. Απλά δράταμε με τις ευκαιρίες όπου συναντιόνται τρεις θεσμοί για να συζητήσουν για το θέμα αυτό και επιθυμώ να απευθυνθώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλώντας το να υποστηρίξει ανεπιφύλακτα τις προτάσεις της Επιτροπής γιατί αυτό θα είναι ένα σαφές μήνυμα για το Συμβούλιο της Δευτέρας γνωρίζουμε ότι ορισμένα κρατημέλη έχουν ακόμα να κάνουν κάποια βήματα πριν δείξουν ότι συμφωνούν το όντι με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλύτερη θα είναι σήμερα η απόφαση του Κοινοβουλίου, τόσο καλύτερα θα είμαστε προετοιμασμένοι για τη Δευτέρα. Γιατί υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν αυταπατώμενοι ότι κλείνοντας τα σύνορα και στέλνοντας όλους αυτούς τους ανθρώπους πίσω ότι έτσι μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Και υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι απλά ανοίγοντας όλα τα σύνορα και αφήνοντας όλους να εισέλθουν ότι μπορούμε έτσι δήθεν να λύσουμε το πρόβλημα. Λυπάμαι πάρα πολύ, όπως είπα αυτά είναι αυταπάτες. Ε, οι προτάσεις μας ε, πρέπει να είναι σαφείς και υπάρχει και κάτι άλλο, ότι αυτά μπορεί να μοιάζουν απλά, υπάρχει όμως το μειονέκτημα ότι δεν είναι εφαρμόσιμα. Γιατί το να κλείσει κανείς τα σύνορα απλά σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε τις ε, πλέον θεμελιώδεις αξίες μας των Ευρωπαίων και σημαίνει επίσης ότι δρούμε ξεκάθαρα παραβιάζοντας τις νομικές μας υποχρεώσεις. Ανοίγοντας τα σύνορα και αφήνοντας όλους να εισέλθουν, αυτό βέβαια θα σημαίνει ότι ε, λέμε τέλος ε, στο κοινωνικό μοντέλο ως το γνωρίζουμε σήμερα γιατί δεν μπορούμε να στηρίξουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ως εκ τούτου οφείλουμε να προβούμε σε σαφή διαχωρισμό ανάμεσα σε εκείνους που τους αξίζει η αλληλεγγύη μας γιατί φεύγουν διοκόμενοι και διαχωρισμός από τους άλλους που επιθυμούν να έχουν ένα καλύτερο μέλλον, αλλά δεν πρέπει να κάνουν κατάχρηση του δικαιώματος ασύλου για να επιτύχουν το στόχο τους. Ως εκ τούτου πρέπει να υπάρχει συνδυασμός ανάμεσα στην αλληλεγγύη και την ευθύνη. Αλληλεγγύη με εκείνους που χρειάζονται καταφύγιο. Αλληλεγγύη από πλευράς εκείνων των ε, κρατών ε, που κοντεύουν σχεδόν να σκάσουν ε, γιατί είναι εκείνοι που δέχονται την πρώτη φουρνιά των μεταναστών. Είναι απαραίτητο να υπάρχει αλληλεγγύη με αυτά τα κράτη. Αλληλεγγύη βέβαια και με τους μετανάστες και με τα κράτη αυτή της Ευρώπης που τη χρειάζονται σήμερα. Αυτή είναι η βάση των προτάσεών μας, αλλά επιτρέψτε μου παράλληλα να απευθύνω έκκληση και για υπευθυνότητα. Να υπάρχει καλύτερη φύλαξη των συνόρων μας. Να γίνεται ταχύτατη καταγραφή όσων φτάνουν στα σύνορα για να μπορούμε ακριβώς να κάνουμε αυτή τη διαφοροποίηση των εχόντων δικαίωμα ασύλου και των άλλων που δεν έχουν. Με τον τρόπο αυτό αυτοί που δεν έχουν δικαίωμα θα μπορούμε να τους επαναπέμψουμε ταχύτατα. Να υπάρχει υπευθυνότητα όσον αφορά την οργάνωση της ε, πρώτης αποδοχής ε, των προσφύγων. Όλα αυτά τα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω και να δώσω μετά το λόγο στη Φεντερίκα. Αυτό που κάνουμε σήμερα και αυτό που θα κάνουμε τη Δευτέρα μεθαύριο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη μοίρα της Ευρώπης. Όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με τη μοίρα της Ευρώπης ως μια κοινότητα αξιών όπου καλούμεθα να δείχνουμε σεβασμό ε, να υποκλεινόμεθα σε αυτό που δείχνουν σήμερα άριθμοι Ευρωπαίοι πολίτες. Δηλαδή μια ανθρωπιά, ανθρωπιά που με κάνει εμένα τόσο υπερήφανο που είμαι Ευρωπαίος. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ τον Αντιπρόεδρο κύριο Τίμερμανς και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην ύπατη εκπρόσωπο την κυρία Φεντερίνη. Μογκερίνη, με συγχωρείτε, Φεντερίκα Μογκερίνη. Σα ευχαριστώ πολύ. Είναι οριστική αυτή η στιγμή και θα ορίσει την ένωση μας. Η... Τα λόγια είναι σημαντικά, πιστεύω, και η κρίση των προσφύγων που αντιμετωπίζουμε όχι μόνο εμεί, αλλά όλη η περιοχή, όλη η περιφερειά μας, νομίζω ότι κλονίζει και βάζει σε μια δοκιμασία τις αξίες μας. Είναι η στιγμή τη αλήθεια. να δούμε αν είμαστε πραγματικά Ευρωπαίοι και αν είμαστε πραγματικά Ένωση. Αυτά. η ευθύνη μας να προασπιστούμε, να υπερασπιστούμε τα, τις ζωές των ανθρώπων και τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και προς αυτούς που είναι σε κατάσταση ανάγκης. Αλλά είναι μια δοκιμασία και για την διεθνή αξιοπιστία μας, ξέρετε. Μην πιστεύετε ότι μπορούμε να κυκλοφορούμε σε όλο τον κόσμο και να προασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα εάν δεν εφαρμόσουμε τα πιο υψηλά πρότυπα για το άσυλο μέσα στην Ένωση. Don't think... Μην πιστέψετε ούτε να σας περάσει από το μυαλό ότι μπορούμε να προωθούμε όλα αυτά και τη συνεργασία μεταξύ των μελών που είναι σε ένα σύραξη στην παρούσα φάση, αν δεν αποδεχτούμε τους άλλους μέσα στις ίδιες μας τις κοινωνίες και δεν μπορέσουμε εμείς οι ίδιοι να βρούμε την ενότητα. Η εξωτερική μας αξιοπιστία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενιαία συνεκτικότητά μας. Μην φανταστείτε ότι είναι μόνο η εξωτερική αντίδραση στην κρίση αυτή. Όπως δεν μπορεί να υπάρξει μόνο εσωτερική αντίδραση στην κρίση και οι δύο διαστάσεις των δράσεών μας, της ταυτότητάς μας, μπορούν να ενδυναμωθούν ή να αποδυναμωθούν. Και είναι αλληλένδετε. Αυτή είναι η να αποδυναμωθουν και ειναι αλληλενδετες αυτη ειναι η αληθεια Δεν μα αρέσει είτε όχι. Για να είμαστε λοιπόν αξιόπιστοι, δεν αρκούν αυτά που κάνουμε. Θα πρέπει να δράσουμε γρήγορα αποτελεσματικά και ενωμένοι. Σήμερα μία ανακοίνωση ε, προλιάνει το έδαφος για τις αντιδράσεις που χρειάζονται για την κρίση αυτή. Όλοι ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κάποια μαγική λύση, γρήγορη λύση, εύκολη λύση για την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε και πιο πολλές δράσεις θα αποδώσουν καρπούς μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ωστόσο είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε τώρα. Το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το εξηγήσουν αυτό οι πολιτικοί ποιος είναι ο λόγος που θα, κάνουμε, θα λάβουμε δράσεις οι οποίες θα αποδώσουν καρπού σε χρόνια σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά αν δεν το κάνουμε αυτό υπεύθυνα, οι επόμενες γενιές θα έρχονται συνέχεια αντιμέτωπες με τα ίδια προβλήματα. Η εξωτερική δράση λοιπόν για πρώτη φορά επίσης μας βρίσκει ενωμένου. Θα πρέπει να έχουμε και εσωτερική ενότητα όμως για τις εσωτερικές πολιτικές. Είναι απαραίτητο φυσικά αυτό για τις δράσεις μας. Πρώτη προτεραιότητα, να σώσουμε ζωές. Ο Πρόεδρος ε, παρουσίασε το πόσο μεγάλες προσπάθειες γίνονται σε, αυτή την, ε, σε αυτό το τομέα και πόσες ζωές έχουν ε, γλιτώσει. Να αντιμετωπίσουμε επίσης κατά δεύτερον τις αιτίες, κατά τρίτον να καταπολεμήσουμε τους διακινητές. Όχι μόνο στη θάλασσα, παντού. Γιατί είναι θέμα ασφάλειας αυτό, γιατί οι οικονομικές ε, ροές και τα έσοδα μπορούν να χρηματοδοτήσουν οποιαδήποτε διαδικασία, οποιαδήποτε δραστηριότητα. Η στρατηγική μας ήταν συνεκτική από την αρχή της ε, πολιτικής μας δράσης. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε μόνο το τελευταίο κομμάτι της, της τραγωδίας. Πρέπει να κοιτάξουμε όλα τα βήματα της Οδύσσιας των προσφύγων. Οι πιο πολλοί που έρχονται στην Ευρώπη σήμερα αυτό θα πρέπει να κοιτάξουμε καταρχά. Τέσσερα εκατομμύρια έχουν φύγει από τη Συρία. Μεταξύ Συρία και Ιράκ, πάνω από 10 εκατομμύρια έχουν φύγει από τα σπίτια του και είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι. Να διευκρινίσω το εξή. Του τελευταίου μήνε έχουμε εστιαστεί και καλά κάναμε στου ε, μειονοτητέ ε, στην ε, Μέση Ανατολή, στου ε, χριστιανού, Ισίτε και του καθεξή, για να υποστηρίξουμε τα δικαιώματά του να επανέλθουν, να ξαναπάνε στι κοινότητε που ζουν εδώ και αιώνε. Αλλά να πω και με πάσα σαφένεια ότι δεν μπορούμε να τις προστατέψουμε μόνο όταν είναι μακριά μας. Έχουμε καθήκον να τις προστατεύουμε όταν μας προσεγγίζουν κιόλας και είναι πιο κοντά μας. Μακροπρόθεσμη απάντηση προφανώς είναι να μπει ένα τέλος στους πολέμους και στις συγκρούσεις γιατί αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα ε, του ολοκαυτώματος και Ισλαμικού κράτου και θα πρέπει να κοιτάξουμε όλε τι νέε ευκαιρίε. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τον πόλεμο, τι γίνεται με τη συνεργασία με όλε τι ε, περιφερειακέ δυνάμει και έχουν ξεκινήσει εργασίε προ την κατεύθυνση αυτή. Κατά δεύτερον, η συνεργασία με την ε, διεθνή κοινότητα, με τι υπηρεσίε του ΟΗΕ, με τι χώρε προέλευση και διακίνηση και με αυτέ που παράγουν ένα ε, εντυπωσιακό αριθμό προσφύγων έχουμε κινητοποιήσει 4 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσουμε τους εσωτερικά εκτοπισμένους ε, στη Συρία, στην Τουρκία, στο Λίβανο και στο Ιράκ. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση, η Λιβύη. Δεν είναι χώρα προέλευσης, αλλά χώρα διακίνησης. Ε, ένας ανοιχτός διάδρομος θα έλεγα. Κάνουμε λοιπόν ε, νύχθημερών προσπάθειες για να μπορέσουμε να πετύχουμε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας στη Λιβύη που θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την κυβέρνηση εσωτέρων για να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον ανοιχτό διάδρομο διέλευση. Να σα πω ότι εργαζόμαστε πολύ σκληρά προ την κατεύθυνση αυτή, αλλά κοιτάμε και τον νότο τη Λιβύη. Αν εστιαστούμε μόνο στα θαλάσσια σύνορα τη Λιβύη, ξεχνώντα τι γίνεται με τα χερσαία σύνορα, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε το θέμα αυτό του διαδρόμου. Και γι' αυτό λοιπόν ξεκίνησα ένα διάλογο άνευ προηγουμένου με τις χώρες Σαχέλ και με τον Νιγηρά ιδιαίτερος, αλλά όχι μόνο με τον Νιγηρά. Και όπως ξέρετε σήμερα καταθέτουμε την πρόταση για ένα καταπίστευμα για την Αφρική για να προωθηθούν οι οικονομικές ευκαιρίες, η ανάπτυξη, η ασφάλεια, καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης με ένα καθεστώς ίσης εταιρικής σχέσης με τους Αφρικάνους εταίρους όργανα θα δώσουν 1,8 δισεκατομμύρια στο ταμείο αυτό. Και αναμένω από όλα τα κράτη-μέλη να κάνουν το μερίδιο από τι αναλογίε. Δεν μπορούμε να ζητάμε προσπάθειε από ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά να μην δίνουμε λεφτά. Να το θυμηθείτε όταν θα συζητήσουμε τον προπολογισμό. Θα πρέπει να υπάρξει μια συνεπτική αντίδραση και σε ό,τι αφορά τη λήψη των αποφάσεων. Ένα περιφερειακό καταπίστευμα για τη Συρία έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία τους τελευταίους μήνες και το, πρώτη σύμβαση που έχει τέτοια εφαρμογή αφορά την ε, εκπαίδευση και τα σχολεία. Επειδή πιστεύουμε ότι η Συρία θα χάσει μια ολόκληρη γενιά λόγω του πολέμου και της ε, εξορίας, θα πρέπει να επενδύσουμε στα παιδιά για το μέλλον της ε, και την ασφάλεια της περιοχής, αλλά και για το δικό μας το μέλλον, γιατί δική μας την ασφάλεια, γιατί είναι Ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε κατά της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά τους διακινητές. Ε, συνεργαζόμαστε και με τις χώρες διέλευσης και εστιαζόμαστε αντιδρά στην Μεσόγειο. Οι ναυτικές μας επιχειρήσεις στη Μεσόγειο έχουν πλέον ε, εκπληρώσει τους στόχους της πρώτης φάσης σε ό,τι αφορά τις διατρόπους των διακινητών, τα χρηματικά του χρηματικού πόρου που έχουν και τι μεθόδου. Σε πέντε εβδομάδες, σε 16 περιπτώσει θα μπορούσαμε να έχουμε ε, πιάσει του διακινητέ και να τους προσφάγουμε στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό στο Λουξεμβούργο την προηγούμενη εβδομάδα με τους υπουργούς τους αρμόδιους συμφωνήσαμε να περάσουμε στη δεύτερη φάση στη, στα ανοιχτό πέλαγος και ζητούμε λοιπόν από τα κρατημέλη να συμβάλλουν με πόρους στην αποστολή αυτή, γιατί πιστεύω ότι αυτό αποτελεί επίσης μια ευκαιρία να επιδείξουμε ότι όπου υπάρχει πολιτική βούληση, ενότητα και αίσθηση κατεπήγοντος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα στρατιωτικά μέσα τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας. Αλλά έχω και κάτι άλλο για το οποίο είμαι πολύ υπερήφανη. Αυτές τις πρώτες εβδομάδες της κοινή δράση στη Μεσόγειο σώσαμε 1500 ζωές γυναικών και ανδρών στη θάλασσα. Αυτός δεν είναι ο βασικός στόχος της ε, αποστολής, αλλά αποτελεί πολύ σημαντικό ε, στοιχείο. Το Νοέμβριο θα γίνει σύνοδος για την μετανάστευση, όπου θα συγκεντρωθούν Ευρωπαίοι ηγέτες και Αφρικανοί ηγέτες και στην διαδικασία Χαρτούμ και Ραμπάτ και της Αφρικανικής Ένωσης και τα κράτη της, ε, των Δυτικών Βαλνίων θα γίνει η διάσκεψη για τον διάδρομο των Δυτικών Βαλκανίων και τα δύο θα πρέπει λοιπόν να τα προσέξουμε εξίσου αυτό θα φέρει από κοινού και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, και την Τουρκία και τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων. Και κλείνοντας να πω ότι δεν είναι αυτή η εποχή, η εποχή για συστηματισμούς. Αυτό είναι το εύκολο ως πολιτική, για να τα πω μα, δεν μας ζητούν συναισθήματα να εκφράσουμε, όχι αποφάσεις καλούμαστε να πάρουμε οι οποίες συνάδουν με τα συναισθήματά μας και να επιμείνουμε και ισχυροί σε αυτά. Δεν φτάνουν τα συναισθήματα. Και σε αυτή την χρονική στιγμή βρισκόμαστε λοιπόν. Ελπίζω λοιπόν ότι όλα τα θεσμικά όργανα και η κοινή γνώμη, γιατί το συνέστημα, ξέρετε, επηρεάζει την κοινή γνώμη, αλλά αυτό μπορεί εύκολα να αλλάξει, να το ξέρουμε αυτό. Θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Να αλθούμε στο ύψος των περιστάσεων και στις προκλήσεις σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές τις οποίες ε, μας έχει επιφυλάξει η πρόσφατη ιστορία μας και αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μόνο οι ζωέ των ανθρώπων και αυτά είναι η ζωή ενός ανθρώπου και μόνο, αλλά και η κατάσταση της ένωσής μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μογκερίνη και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Παραμόπουλο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως παρατηρήσατε, η ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης έφερε ως επιτοπλίστων επί του μεταναστευτικού ζητήματος και μας δείχνει ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Ο πρόεδρος ήταν ξεκάθαρος και το ίδιο θέλω κι εγώ. Θέλω να είμαι σαφής. Η διαχείριση της ε, μετανάστευσης είναι κράστες, είναι δοκιμή αν θέλετε για την, ε, και λιδία λίθος για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Φραν Τίμερμαν και τη Φεντερίκα Μοκερίνη για τι εναρκτήριε παρατηρήσει του, αλλά και για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε του περασμένου μήνε ε, κατά την σύσταση αυτού του φιλόδοξου πακέτου που τόσο χρειαζόμαστε. Το σημερινό πακέτο είναι η απάντηση που δίνουμε σε μια προσφυγική κρίση ανεφροηγουμένου που ε, συμβαίνει και εκτελήσεται ακριβώς μπροστά στα μάτια μας. Και όσο διωγγώνεται αυτή η κρίση, τόσο, πρέπει, τόσο πιο θαραλέες και σφαιρικές πρέπει να είναι οι απαντήσεις μας, τόσο πιο φιλόδοξη πρέπει να είναι η απάντηση που δίνουμε. Αυτή είναι η Ευρώπη που θέλουμε, αυτή είναι η Ευρώπη που πρέπει να έχουμε. Σήμερα λοιπόν εισηγούμαστε τέσσερα πολύ συγκεκριμένα μέτρα που μέσω μακροπρόθεσμα θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε το σύνολο των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας. Η σημαντική αύξηση των αφήξεων μετά το καλοκαίρι είναι κάτι που δεν μπορούν τα κράτη-μέλη εισόδου να αντιμετωπίσουν από μόνα τους. Για να διαχειριστούμε αυτό το ζήτημα χρειαζόμαστε μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση και γι' αυτό τώρα προτείνουμε να επανεγκαταστήσουμε 120.000 ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη δίωξη, από την καταστολή, από το χάος, από τον πόλεμο, από την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ουγγαρία, βάσει μιας κλίδας κατανομής. Αυτή η νέα πρόταση προστίθεται στα μέτρα που καταθέσαμε πριν από το καλοκαίρι για την μετεγκατάσταση 40.000 ατόμων από την Ιταλία και από την Ελλάδα περιμένουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα υπερψηφίσουν αργότερα τη νέα πρόταση και μελλοντικά θα υποστηρίξουν, υποστηρίξουν συγγνώμη, και το προσωρινό καθεστώς με την κατάσταση. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αντλήσουμε τα διδάγματα από την τωρινή κρίση. Η Ευρώπη δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένη για να αντιμετωπίζει ξαφνικές και μαζικές προσφυγικές ροές. Χρειαζόμαστε σε διαρθρωτικού τύπου λύσεις στο μέλλον, τόσο ώστε με συστηματικό τρόπο να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη και να εξασφαλίσουμε προστασία για αυτούς που πραγματικά τη χρειάζονται. Και γι' αυτό προτείνουμε σύσθεση ενός μονίμου μηχανισμού ε, την κατάσταση τροποποιώντας τον κανονισμό Δουβλίνου. Ταυτόχρονα, Αυξάνοντα την υποστήριξή μα για τη στέγαση αυτών που χρειάζονται διεθνή προστασία, θα πρέπει να φροντίσουμε ούτω ώστε αυτοί που δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αμελητοί να, να επιστρέψουν. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για τα κράτη-μέλη, δηλαδή σταθερά θα πρέπει να επεξεργάζονται μη τεκμηριωμένα τέτοια αιτήματα τα κράτη-μέλη, ούτω ώστε τους ανθρώπινου και του οικονομικούς του πόρου να μπορέσουν να τους διοικητεύσουν σε θεμητά αιτήματα. Αυτοί που, ε, για αυτούς που χρειάζονται κατεπηγόντως διεθνή προστασία. Και γι' αυτό σήμερα προτείνουμε την εισαγωγή μιας ε, λίστας ασφαλών χωρών, ε, συμπεριλαμβανομένων και των Βαλκανικών χωρών και της Τουρκίας. Το 2014 οι πήκοοι από αυτές τις χώρες κατέθεσαν πάνω 17% ε, των 560.000 αιτήσεων που εξετάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα αιτήματα συνεπάγονται ένα πολύ σημαντικό άχθος για το σύστημα σύλλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι η συντριπτική πλειοψηφία ε, ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ήταν στοιχειοθετημένη. Η εξέταση των ετοιμάτων για παροχή ε, διεθνούς προστασίας θα επισπευστεί βάσει του νέου συστήματος ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα του συστήματος ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτρέποντας τα κράτη-μέλη να διοχετεύουν τους πόρους αυτούς που χρειάζονται την προστασία και να επιστρέφουν ε, στις χώρες τους ταχύτερα όσους δεν δικαιούνται αυτή την προστασία. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαμηλότατο ποσοστό επιστροφών και ε, αυτό φτάνει το 40% για τους ε, υπηκούς τρίτων χωρών. Όπερ και υπονομεύει την αξιοπιστία της μεταναστευτικής μας πολιτικής και γι' αυτό σήμερα παρουσιάζουμε και ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιστροφής, ούτως ώστε να ε, είναι ξεκάθαρη πλέον η πολιτική επιστροφών. Είναι σήμερα μια ευκαιρία για μα ε, να εισηγηθούμε μια σειρά δράσεων, ώστε σε επιχειρησιακό επίπεδο να ενισχυθεί η συνεργασία των κρατών μελών ε, και να χρησιμοποιήσουμε τη μόχλευση των διμερών μας σχέσεων, ακόμη και σε εξωτερικές μας σχέσεις, για την επανεγκατάσταση των υπηκών τους. Σας υπολογίζουμε στη δική σας βοήθεια για την εφαρμογή αυτού του πακέτου, όπως ακριβώς το κάνατε και παρεμπιπτόντως να σας συγχαρώ και πάλι, ε, για το προηγούμενο πακέτο μας υποστηρίξατε στην απαρχή της προσπάθειάς μας ε, για να συστήσουμε μια κοινή ε, μεταναστευτική πολιτική. Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω και πάλι και υπολογίζω στη βοήθειά σας σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Αβραμόπουλε. Θα έχουμε την ε, χαρά να σε ακούσουμε και σε δευτερολογία. Πρώτα θα μιλήσουν οι αρχηγοί των πολιτικών ομάδων. Και θέλω απλά να σε επισημάνω ότι έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Ε, εντάξει, θα είμαι λίγο εμπέληκτος όσον αφορά το χρόνο, αλλά δεν θα δεχτούμε μπλε κάρτες. Και όσον αφορά τη διαδικασία Catch the Eye θα δούμε κατά πόσον θα μπορέσουμε να κερδίσουμε λιγάκι χρόνο. Γιατί στις, ε, στη μια μισή ώρα πρέπει να ψηφίσουμε για σημαντικές εκθέσεις. Το λόγο έχει ε, το ΕΛΚ ο κύριος Κερσία Ντεγκουέρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Υπάρχουν ε, άνθρωποι που ε, ρισκάρουν τη ζωή τους ε, για να ξεφύγουν από την βία του Ισλαμικού κράτους. Πρόκειται για πρόσφυγες, πρόκειται για ανθρώπους που πρέπει να βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλωσορίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι αποφασιστική σημασία και πρέπει κατεπηγόντως να εγκριθεί αυτή η πρόταση, διότι το φαινόμενο αυτό θα παρατηρείται για πάρα πολύ καιρό. Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν πάγιο δεσμευτικό κοινό μηχανισμό δυνάμει του άρθρου 47.2 της συνθήκης με τρόπο ώστε να υποδεχόμαστε με αξιοπρεπή τρόπο τους πρόσφυγες. Όλοι θα πρέπει να επιδείξουν αλληλεγγύη, όλα τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς που χρειάζονται τη βοήθειά μας σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα των αδυνάτων. θα πρέπει να οριοθετήσουμε σωστά το φαινόμενο ώστε να καταπολεμήσουμε και την τρομοκρατία και την βία ε, του Ισλαμικού κράτους ε, και των θεσμών του θα πρέπει να ε, επιτεθούμε σε αυτό το κακό στη ρίζα του και να συνεχίσουμε τη δράση που αρχίσαμε το 2012. Κύριος Πιτέλα, εκ μέρου των Σοσιαλιστών, τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Σασόλη. Ε, κύριε Υπουργέ Σμιτ, κύριε Αντιπρόεδρη ε, Τίμερμαν ε, και Μογκερίνη, Κύριε Επίτροπε, κύριε Αβραμοπούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που έχετε κάνει. Ε, θέλω να επισημάνω ότι η δική μου η πολιτική ομάδα, της οποίας προείσταμε, είναι εκείνη που εξέφρασε και κατέθεσε αρκετές προτάσεις από αυτές ε, τις οποίες ανέφερε σήμερα και ο κύριος Αβραμόπουλος στο πακέτο μέτρων που πρόκειται να ληφθεί. Θέλω να πω το εξή ότι όσον αφορά τη μετανάστευση δεν είναι δυνατόν να ε, γύρουμε τύχη στη θάλασσα. Δεν είναι δυνατόν να συγκρατήσουμε ανθρώπους που θέλουν να ξεφύγουν από τον πόλεμο. Μα τι είναι αυτά, τι συζητάμε εδώ. Αυτά είναι μόνο λόγια που λέγονται για ε, σκοπούς προπαγάνδας. Πιστεύει κανείς άραγε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να λυθεί το πρόβλημα των ε, προσφύγων και των μεταναστών. Μα εγώ θεωρώ ότι αστευόμαστε. Αυτό είναι καθαρά κομματική προπαγάνδα για να κερδίσει κανείς ψήφους. Πρέπει να είμαστε σοβαροί προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σοβαρές προτάσεις που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα έκτακτης ανάγκης, αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Οι προτάσεις ε, προβλέπουν ένα μόνιμο σύστημα το οποίο θα μπορεί να δραστηριοποιηθεί οποτεδήποτε προκύψουν παρεμφερείς κρίσεις. Γιατί θα προκύψουν τέτοιου είδους κρίσεις. Βεβαίως υπάρχει και το θέμα των οικονομικών μεταναστών και αυτό καλούμεθα να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρό τρόπο, να κατανοήσουμε ποιες είναι οι ανάγκες της ε, κοινωνίας και της ε, αγοράς εργασίας των κρατών μελών, σίγουρα να γίνονται έλεγχοι με κοινού ε, κανόνες ε, και κατά την ίδια χρονική στιγμή και προβλέποντας ε, το ίδιο χρονικό διάστημα. Όχι η μία χώρα να θέλει ένα μήνα και η άλλη έξι μήνες για να διαπιστώσει αν τελικά θα γίνει αποδεκτός ο οικονομικός μετανάστης ή όχι. Αναφέρθηκε προηγουμένως η Αφρική και επανήλθε σήμερα η κυρία Μογκερίνη αλλά και ο κύριος ε, Τίμερμαν στην Αφρική. Ξέρετε, η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σημαντική για να ε, καταλήξουμε στο τι θέλουμε να κάνουμε με τη Λιβύη, με τη Συρία. Αυτά είναι κράτη μη κράτη. Από εκεί φεύγουν οι άνθρωποι. Μα τι να κάνουν άλλο. Και εμεί αν ήμασταν στη θέση του και εμεί θα ξεφεύγαμε. Θα θέλαμε να καταλήψουμε τη χώρα. Άρα δηλαδή χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη στρατηγική, χωρί δημαγωγικά στοιχεία, με ρεαλισμό, με σοβαρότητα. Απευθύνω λοιπόν τώρα για άλλη μια φορά στο Συμβούλιο γνωρίζω πολύ καλά τη στράτευση του Υπουργού από το Λουξεμβούργο. Θα ήθελα όμως η στράτευση του αυτή, η ευαισθησία του να χαρακτηρίζει το σύνολο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πιτέλα, λέει ο Πρόεδρος. Το λόγο έχει ο κύριος ε, Στίβενς για ένα λεπτό εκ μέρους πολιτικής ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Η κυρία Στίβενς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι πρόσφυγες οι οποίοι μπαίνουν από την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διωχθούν από τη θάλασσα στην Τουρκία και σύμφωνα με την ε, διεθνές δίκαιο απαγορεύεται να επιστρέψει κάποιος σε ε, λιμένα που δεν είναι ασφαλής. Ε, το ΕΝΔΑ θεωρεί ότι είναι ασφαλής χώρα η Τουρκία και σε περίπτωση που δεν είναι κάτι τέτοιο θα πρέπει να αποφανθούν ε, οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν όμως ε, τέτοιες αποφάσεις. Ε. Κοιτάμε μόνο την επιστροφή μέσω της Ιταλίας στη Λιβύη. Η κατάσταση είναι διαφορετική. Ο πρόεδρος Γιούγκερ είπε ότι η Τουρκία είναι υποψήφιο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα ασφαλές κράτος. Αν δεν ήταν ασφαλές δεν θα ήταν ε, κράτος υποψήφιο προστάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Βίκστρομ, επόμενος ομιλητής για δύο λεπτά, ε, δυόμιση λεπτά εκ μέρους της, των φιλελευθέρων. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τι τελευταίε δύο εβδομάδε ε, το θέμα των προσφύγων έχει λάβει ένα όνομα αν θέλετε, μία ιστορία, με μία εικόνα. Καταλάβαμε ότι πίσω από κάθε πρόσφυγα είναι όνειρα, είναι φιλοδοξίες, είναι μια οικογένεια που μένει πίσω. Είναι λοιπόν θέμα αξιοπρέπειας, ευρωπαϊκής αξιοπρέπειας που βρίσκεται στις τουρκικές ε, ακτές μαζί με τον Αλαντούλη, ο οποίος βρίσκεται άψυχος έχασε τη ζωή του, αλλά έφερε πάθος και ε, συμπόνια στην ευρωπαϊκή συζήτηση για την ε, προσφυγιά και τη μετανάστευση. Γι' αυτό λοιπόν θα τον θυμόμαστε για πολύ καιρό μετά τις πρόσφατες τραγωδίες. Αισθάνομαι περηφάνεια όταν βλέπω πολίτες σε όλη την Ευρώπη να βγαίνουν στους δρόμους για να υποδεχτούν τους πρόσφυγες της κοινωνίας τους. Γιατί κύριε Πρόεδρε, αυτοί έχουν δείξει πολύ πιο πολύ ανθρωπιά και ραχοκοκαλιά τις τελευταίες εβδομάδες από τους πιο πολλούς πολιτικούς τις τελευταίες δεκαετίες μάλιστα. Οι πολίτες μας δείχνουν τι σημαίνει η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές αξίες και τι μπορεί να σημαίνει στην καλύτερη εκδοχή της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εξακολουθούμε να ακούμε κάποιες φωνές μεταξύ των ηγετών των κρατών μελών που παραπονιούνται για τους ε, παράνομους μετανάστες. Και πρέπει να σας πω κύριε Πρόεδρε ότι με έχει κουράσει πια αυτή η ρητορική. Πώς ε, να μπει δηλαδή κάποιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν φεύγει από καθεστώς πολέμου και να ζητήσει άσυλο αφού δεν επιτρέπουμε να ζητείτε άσυλο στις ε, πρεσβείες και στα προξενίες μας. Εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να καταρτήσουμε μια νομοθεσία για τους ε, μεταφορείς ε, που θα επιτρέψουν στα άτομα που θα μπορούν να μπαίνουν στα αεροπλάνα. Εμείς λοιπόν δημιουργήσαμε αυτό το φαύλο κύκλο. Εμείς θα πρέπει να τον αλλάξουμε. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την πολιτική για το άσυλο στην Ευρώπη, να την προσαρμέσουμε στον αιώνα μας για να δώσουμε ασφαλείς οδούς. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε για δεσμευτικές ποσοστώσεις για τους μετανάστες. Και φυσικά είμαστε υπέρ των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την ομάδα μας. Είναι καθοριστική η στιγμή για την Ευρώπη και περιμένουμε μια καλύτερη ημέρα. Παρόλα, Το λόγο λοιπόν έχει τώρα εκ μέρου ε, τη Ενωμένη ε, Αριστερά ε, ο κ. η κυρία Σμάν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Τέσσερα εκατομμύρια πρόσφυγε από τη Συρία 4 εκατομμύρια από το Ιράκ, 3,5 από το Αφγανιστάν, 2,5 εκατομμύρια από τη Λιβύη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των πολέμων, των πολέμων στο Ιράκ, του Αφγανιστάν και η υποστήριξη της Λιβύης. Υποστήριξαν με όπλα τον πόλεμο στη Συρία. Και όταν φτάνουν στο κατόφλι μας οι πρόσφυγες, τι κάνουμε, προσπαθούμε να βρούμε νομικές λύσεις, κάποιον κανονικό ανθρωπιστικό διάδρομο, ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Όχι, όχι και όχι. Προστασία, ούτε αυτό. Τι κάνουμε. Ο Λάντε μελετά την κατάσταση του Ισλαμικού κράτους στην ε, Συρία. Ο Κάμερον προσπαθεί κάτι να κάνει στη Συρία. Ο Μωράιο προσπαθεί να προβεί σε στρατιωτικές παρεμβάσεις στην Συρία. Ο αιτία είναι ο πόλεμος και η λύση δεν είναι στις βόμβες. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σαρτζεντίνη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο πρόεδρος Γιούγκερ είπε σήμερα το πρωί στην ε, δήλωση για την κατάσταση της Ένωσης ότι το, η εργασία σημαίνει ε, αξιοπρέπεια. Θα πρέπει να επιτρέπουμε να εργάζονται οι πρόσφυγες από τη στιγμή που μπαίνουν στην Ένωση. Και είπε επίσης ο Πρόεδρος ότι θα πρέπει να επιτρέψουμε και την μετανάστευση. Οικονομική μετανάστευση, μετανάστευση των εργαζομένων, γιατί είπε στη συνέχεια ότι δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση αν δεν υπάρχουν άλλες μορφές ε, ε, μετανάστευση. Ρωτώ τον κύριο Βραμόπουλο και τον κύριο Τίμερμαντ. Οι προτάσει που κάνουν τώρα είναι καλέ και στεναρέ. Αλλά το επόμενο βήμα το επόμενο βήμα που ανακοίνωσε ο κύριος Γιούγκερ για την ε, μετανάστευση εργασίας δεν πρέπει να περιμένει, γιατί όντως το να εργάζεται κανείς σημαίνει το να έχει αξιοπρέπεια. αξιοπρέπεια. Αυτό λοιπόν ελπίζω να μπει επιτάπητος πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Κοράο, εκ μέρους της ομάδας EFD, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εμείς συνεχίζουμε να μιλάμε για έκτακτη ανάγκη. Είναι βέβαια σαφές ότι δεν μπορεί να είναι έκτακτη ανάγκη κάτι που συνεχίζεται για χρόνια. Εμείς πιστεύουμε ότι ε, βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρωτοφανή έξοδο, ε, αποτέλεσμα μιας ε, πολιτικής εκμετάλλευσης στις χώρες από τις οποίες φεύγουν οι άνθρωποι. Μένεται ο πόλεμος. Εμείς λοιπόν τοποθετηθήκαμε Καταλήξαμε σε ένα σύνθημα και το προβάλλουμε και σήμερα. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που μπορούν να δραστηριοποιηθούν, αλλά αυτά υποκρίνονται διότι τα κρατημέλη είναι εκείνα τα οποία στο όνομα των δικών τους των οικονομικών συμφερόντων και του νεοφιλελευθερισμού δεν κάνουν τίποτα. Είναι λοιπόν λυπηρό να βλέπει κανείς πρωθυπουργού όπως τον Ιταλό ε, να ε, ζητάνε βοήθεια ε, και να καταφεύγουν σε πολιτικά μέσα έχοντας όμως ξεχάσει ότι υπάρχει αυτό το παιδάκι που σκοτώθηκε αλλά την προηγούμενη μέρα δώσανε όπλα στους Σύριους. Επόμενος, ε, ο κύριος ε, Λίνσκι για ένα λεπτό παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι αυτό που διαπιστώνουμε είναι το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι που χρειάζονται προστασία και βοήθεια θα πρέπει να την χάνουν αυτή τη προστασία και τη βοήθεια. Δεν δείτε θέμα από αυτού, γιατί το μόνο που συζητάμε είναι πού θα τους βοηθήσουμε. Και εδώ υπάρχουν τρία σχέδια. Πρώτον, το σχέδιο της Ενωμένη ΕΕ, Αριστεράς, το σχέδιο των κομμουνιστών και υπάρχει και ένα άλλο σχέδιο. Το δικό σας το σχέδιο είναι να του αφήσει καλείστε όλους να έρθουν εδώ. Δεν ρωτάτε αν είναι πρόσφυγες με βάση τη συνθήκη της Γενέβης, ούτε ρωτάτε αν είναι νόμιμοι μετανάστες, ούτε όμως αν είναι ε, μαχητές του ISIS. Λέτε, ελάτε όλοι εδώ. Εμείς τα πατριωτικά κόμματα λέμε ότι αυτή τη βοήθεια να την προσφέρουμε επιτόπου στα Ισλαμικά κράτη. Εκεί να γίνουν οι μονάδες ε, πρώτης ε, καταγραφής. Να δημιουργήσουμε σαφείς και ασφαλείς ε, ζώνες. Γιατί να μην συμπεριλάβουμε και τα κράτη του κόλπου. Αυτοί να βοηθήσουν τους αδελφούς τους και να εμπλακούν και οι Ηνωμένε Πολιτείε που και αυτές φέρουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στους, από τους μη εγγεγραμμένους. Βόιτ, ε, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα το πρωί άκουσα από το στόμα του κυρίου Γιούγκαρ ότι δεν είμαι Ευρωπαίος, γιατί εγώ δεν έχω πάει ούτε στο σταθμό, ούτε έχω πάει να λεπώ στους μετανάστες καλωσορίσατε. Ξέρετε γιατί δεν το έκανα, γιατί πιστεύω ότι εμείς ε, έχουμε δώσει εντολή εκπροσωπώντας τους ε, λαούς μας να διαφυλαχθεί το δίκαιο και η ταυτότητα των πολιτών μας. Και το ίδιο δικαίωμα ισχύει και έναντι των προσφύγων γιατί και αυτοί που έρχονται εδώ και αυτοί έχουν πατρίδα. Έχουν λοιπόν το δικαίωμα να παραμείνουν στην πατρίδα τους και να διαφυλάξουν τη δική τους την ε, ταυτότητα. Δεν μπορεί κανείς να λύσει τα προβλήματα με το να αφομοιώνει αυτούς τους ανθρώπους. Μα άμα τους αφομοιώσουμε δεν θα επιστρέψουν. Όχι, αυτοί έχουν πατρίδα. Κάποια μέρα να πάνε πίσω στην πατρίδα τους. Εκεί να επενδύσουμε. Στην πατρίδα τους να επενδύσουμε. Εκεί να έχουν μέλος και όχι εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Λέει ο πρόεδρος, η κυρία Μπόζεμπερκ, παρακαλώ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, 260.000 μετανάστες πέρασαν φέτος στην Ελλάδα από τα παράλια της Τουρκίας, ενώ το 2014 77.100 και το 2013 43.000. Το πρόβλημα είναι οξύ και απαιτεί συνεκτική ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Επειδή πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνομοθετεί με το Συμβούλιο, πρέπει να υπάρξει άμεση απόφαση για μόνιμο δεσμευτικό μηχανισμό δίκαιης κατανομής προσφύγων στα κράτη-μέλη, όπως προτείνει η Επιτροπή. Παράλληλα, θα πρέπει οπωσδήποτε η τουρκία να τηρήσει τις συμφωνίες επανεισδοχής που έχει υπογράψει με την ευρωπαϊκή ένωση το 2011 και την ελλάδα τον οκτώβριο του. 2014. τέλος κύριε πρόεδρε μας τιμά το γεγονός ότι η ευρώπη των αξιών στο μεταναστευτικό πρόβλημα δείχνει πάντα το ανθρώπινο πρόσωπό της. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τσίπελ και εσείς παρακαλώ για ένα λεπτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, συνεχώς υποδαβλίζεται αυτός ο φόβος ότι πω, πω, θα έρθουν πάρα πολλοί μετανάστες στην Ευρώπη. Ο κύριος Γιούγκερ Ανέφερε όμως ένα αριθμό, 0,11%. 0,11% είναι αυτό. Και οι περισσότεροι πρόσφυγες εξακολουθούν να έρχονται από χώρε όπως η Συρία και η Ερυθρέα. Οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να ξεφύγουν από διώξεις και από τον πόλεμο. Ε, αυτό όμως ε, το ξεχάσαμε στη σημερινή συζήτηση, συναισθηματικά βέβαια φορτισμένη, γιατί η συζήτηση αυτή είχε ως στόχο να μπουν στο μάτι όλοι οι πρόσφυγες. Και είναι όνειδος ε, το ότι ένα μεγάλο κομμάτι του Συμβουλίου δείχνει να φοβάται μπροστά σε αυτά τα συνθήματα, αντί να υψώσει το αναστημά του και να δείξει αλληλεγγύη και προς τα μέσα και προς τα έξω. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Την επόμενη εβδομάδα πρέπει να δραστηριοποιηθεί το Συμβούλιο και να εφαρμόσει τις επίκαιρες προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτές οι μεγάλες συγκρούσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντα περιέχουν ένα στοιχείο ασφάλειας και ανθρωπιστικής ε, πτυχής. Ο Πούτιν με τους οικονομικούς ε, μετανάστες ε, που έχει προκαλέσει, αυτά έχουν ε, απορροφηθεί από την Πολωνία σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε επιδείξει λεγγύη και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε αυτό σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την ασφάλεια των νότιων συνόρων μας. Ακούσαμε την υπατή αντιπρόσωπο για το τι συμβαίνει και τι δράσεις έχουν αναλυφθεί στην Μεσόγειο, αλλά χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό νέα τοποθέτηση των ατόμων αυτών. Αυτό αναφέρεται στον κανονισμό, αλλά δυστυχώ φοβάμαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδείξει πιο πολύ αλληλεγγύη του ιστορικό της Ένωσης. Για ένα λεπτό, επόμενος ομιλητή. Κύριε Βεριζιά. περίπου 70 εκατομμύρια πρόσφυγοι βρίσκουμε στον κόσμο και 13% στις αναπτυσσόμενες χώρες, μόνο 0,11% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Οπότε πρέπει να κάνουμε τη διαλογή των πραγματικών προσφύγων μας, λένε, ανάλογα με την υπηκότητά τους ή χειρότερα ακόμη. Δεν πρέπει να εξυπηρετούμε μόνο τα δικά μας συμφέροντα κατα... καταρτίζοντας αυτόν τον κατάλογο ασφαλών χωρών. Και τι θα κάνουν αυτοί που χρειάζονται το άσυλο και τι θα γίνουν αυτοί που δεν το δικαιούνται. Θα τους πετάξουμε, θα τους επιστρέψουμε μαζί με τους οικονομικούς μετανάστες, όποια και αν είναι η χώρα προέλευσή τους. Τι μπορούμε να περιμένουμε από το κέρας της Αφρικής και από τις δικτατορίες αυτές ε, στα πλαίσια της διαδικασίας του χαρτού. Με αυτή η διάκριση ανάμεσα στους πραγματικούς πρόσφυγες και τους οικονομικούς μετανάστες ε, θα έχει ως αποτέλεσμα πέσουμε με τα μούτρα σε ένα τείχο. Δεν πρόκειται να δώσουμε λύση διότι θα αυξήσουμε τον αριθμό των θανάτων και βολεύουμε και τους διακινητές οι οποίοι θα κερδοφορήσουν στην πλάτη αυτών των ανθρώπων. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε ε, τις αξίες μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Κέλλερ, ένα λεπτό. Αυτοί συνάδελφοι, η κατάσταση της Ένωσης ε, είναι κάτι που θα πρέπει να μετρήσουμε βάσει τη μεταχείριση που επιφυλάσσουμε σε αυτού που πραγματικά χρειάζονται βοήθεια και δεν είναι σαφή η εικόνα. Ε, ε, υπάρχουν αυτοί που δίνουν, όχι μόνο το τελευταίο Σαββατοκύριακο, αλλά του περασμένου μήνε, τα περασμένα χρόνια και από την άλλη έχουμε κράτη-μέλη που δεν κάνουν τίποτα, που αλληλεκατηγορούνται δεν κάνουν αυτά που θα έπρεπε να κάνουν. Πρέπει να αποφασίσουμε σε ποιο στρατόπεδο ε, θα είμαστε εμεί, σε ποιου θέλουμε να βοηθήσουμε, ποια Ευρώπη θέλουμε να ε, υποστηρίξουμε και να οικοδομήσουμε. Υπάρχουν κάποιοι που μας έδειξαν ναι, ε, το παράδειγμα και δείχνουν ότι άξιζε ε, το Νόμπελ που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κυβερνήσει των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ακολουθήσουν το δρόμο που χάραξαν οι πολίτε. Οι πολίτε μα είναι πολύ πιο προχωρημένοι σε αυτό το τομέα από ό,τι πιστεύουμε. Α ακολουθήσουμε λοιπόν το δρόμο που μα υπέδειξαν τη δική του την πρωτοβουλία. Σα ευχαριστούμε, κύριο Νάταλ. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Αντιπρόεδρε, Επίτροπε, εγώ πιστεύω ότι η απόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό ακολουθεί εντελώς διαφο... Ε, λανθασμένη κατάσταση κατεύθυνση. Εγώ πιστεύω ότι είναι εντελώ ανεύθυνη η Γερμανία και η Σουηδία. Τι θα γίνει αν πούμε ότι όλοι μπορούν να διεκδικήσουν το άσυλο. Μα είναι απλό. Θα έρθουν περισσότεροι, ακόμη περισσότεροι. Θα ε, ρισκάρουν τη ζωή του για να διασχίσουν την Μεσόγειο, το Αιγαίο. Αυτό σημαίνει ακόμη περισσότερα σκάφη, περισσότερου πνιγμού, περισσότερου θανάτου. Και παρότι διαφωνώ εγώ με αυτή την απάντηση που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάθαμε τουλάχιστον κάτι. Το πραγματικό σκάνδαλο εδώ είναι οι χώρε που εμένουν άπρακτες. Και τι εννοώ, ε, τα κράτη του κόλπου, Κατάρ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, ε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και κυρίως αυτοί που, ε, είναι οι σπόνσορες ε, του Ισλαμικού κράτους μιλούν ναι, για την Σαουδική Αραβία. Δεν κάνουν τίποτα. Δεν υποδέχονται κανέναν πρόσφυγα και αυτό που κάνουν είναι να σπρώχνουν τους ομοθρήσκους τους προς την Ευρώπη. Ευχαριστούμε κύριε Νάταλ. Πρέπει να σταματήσετε τα σκάφη, επινοεί ο κύριο Νάταλα Διακόπτεται από τον πρόεδρο Σαλβίνη. Ένα λεπτό. Εγώ άκουσα πολύ υποκριτικές ε, και επικίνδυνες ε, παρεμβάσεις. Αυτό ισχύει για τους Ευρωπαίους, γιατί ξέρετε κάτι. Πρώτα εκείνοι προκαλούν ε, πολέμους και μετά εκπλήσονται που σκοτώνονται παιδιά. Γίνεται λοιπόν εδώ λόγο για business, 150.000 ε, μετανάστες, ε, περίπου 5 εκατομμύρια ε, ευρώ κοστίζουν αυτά στην Ευρώπη, αλλά πάρα πολλοί θεωρούν ότι αυτό είναι business και τρίβουν τα χέρια τους. Ίσως σε αυτή την αίθουσα θα πρέπει να τηρήσουμε ενός λεπτού στη γη, γιατί θα υπάρξουν πάρα πολλοί θάνατοι τους μετανάστες. Κάποιοι λένε ότι υπάρχουν υποπτή για τρομοκρατία κάνουμε ένα λεπτούς υγιή, ε, φοβάμαι ότι αυτό θα πλήξει τη συνείδησή σας. Επίσης θέλω να σας πω ότι χρειαζόμαστε αυτά τα εκατομμύρια τους πρόσφυγες για να διατηρήσουμε τις συντάξεις των Ευρωπαίων. Εσείς ε, πληρώνεστε για να βρείτε κάποια λύση και για τα 25 εκατομμύρια ανέργους στην Ευρώπη. Γκόλνης παρακαλώ για ένα λεπτό. τι βλέπουμε μπροστά μας. Ε, ε, κάποιοι διώκονται και λόγω θρησκευτικών ε, πεπιθήσεων, πολιτικών πεπιθήσεων και προέρχονται από χώρες στον οποίο την αποσταθεροποίηση έχουμε συμβάλει και εμείς και εμείς τους υποδεχόμαστε. Αυτό είναι το φαινόμενο που βλέπουμε ή πρόκειται για μαζική μετανάστευση που μεθοδεύεται σε ανθρωπιστικά προσχήματα. Αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Άκουσα την κυρία Βίξτρομ που μας ε, ε, είπε τα σπαραξικάρδια για το παιδάκι που πέθανε, αλλά συγγνώμη θα ήθελα να τη ρωτήσω γιατί ευθύνονται τα κράτη-μέλη για το θάνατο αυτού του παιδιού που ε, η οικογένειά του ήταν σε ασφάλεια στην Τουρκία. Οι υπεύθυνοι είναι οι Αμερικάνοι και οι, όσοι από τους Ευρωπαίους συνέβαλαν στην αποσταθεροποίηση του Ιράκ και της Συρίας. Ε, είναι τα κράτη του κόλπου ούτε το δαχτυλάκι τους δεν κουνάνε όπως ακούσαμε από το ε, συνάδελφο. Ο αραβικός ε, σύνδεσμος ε, που τίποτα δεν κάνει κατά του Νταές είναι τα κυκλώματα των διακινητών που αναξιοπρεπώς εποφελούνται από, αυτό το, από αυτή τη διακίνηση προσφύγων και εμείς ευθυνόμαστε για όλα. Ο πατέρας αυτού του φτωχού παιδιού που σας πίστεψε είναι αυτός που έχασε. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μέτσολα για λεπτό. Όταν ε, για πρώτη φορά ασχολήθηκα με την πολιτική, με συμβούλευσαν το εξή. Μην μιλά ποτέ όταν έχει εξοργιστεί. Σήμερα όμω δεν θα το κάνω αυτό. Θα μιλήσω. Τα κράτη-μέλη μοιάζουν να συμφωνούν για το πόσα ψάρια μπορούμε να ψαρεύουμε από τι θάλασσέ μα, πόσε πλαστικέ ε, σακούλε ε, να πετάμε. Αλλά όταν όμω τα παιδιά νεκρά βγαίνουν στι ακτέ μα, μοιάζει να μην συμφωνούμε για το τι πρέπει να κάνουμε. Άρα δηλαδή όλα αυτά που λέμε είναι άχρηστα Θέλω επίσης να επισημάνω ότι είμαστε μια ένωση κοινών αξιών, αλλά δεν είμαστε ακόμα μια ένωση κοινών ευθυνών. Και αυτό είναι συλλογική μας αποτυχία. Οι ε, μετανάστες, οι πρόσφυγες ξεφεύγουν από τον πόλεμο, από το θάνατο. Οι πρωθυπουργοί δεν μπορούν να το παραγνωρίζουν. Όλα τα κράτη οφείλουν να εκπληρώνουν την ηθική τους υποχρέωση, να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Τα τείχη και τα φράγματα ε, δεν εξυπηρετούν. Χρειαζόμαστε περισσότερο από εμβαλωματικές λύσεις που εντάξει μας κάνουν να νιώθουμε κάπως καλύτερα πριν όμως η επόμενη κρίση εκθέσει την ανεπάρκειά μας και πράγματι χρειαζόμαστε μηχανισμό ανακατανομής ε, το χρειαζόμαστε ήδη εχθές. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνομαι στους πρωθυπουργού. Αντιμετωπίστε τους δημαγωγούς. Να δείξετε το θάρρος ε, που σημαίνει δώστε ευκαιρία στους ανθρώπους αυτούς και στείλτε ένα σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη είναι στο πλευρό πλευρό εκείνων που δεν έχουν φωνή. Ας γίνουμε το παράδειγμα του κόσμου. Αυτή είναι η πρόκληση της γενιάς μας και δεν πρέπει να μας θυμούνται εκείνους ε, που ε, έδειξαν ητοπάθεια όταν τόσοι πολλοί χτυπούσαν την πόρτα μας. Γιατί εμείς θα είμαστε η γενιά που θα έχει αποτύχει. Επόμενος, ε, Γουαλίν, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ο Σούγκρος ζήτησε το λόγο είναι ιστορική συζήτηση και θα ήθελα να μιλήσω ως Ευρωπαίος. 500 εκατομμύρια πολίτες κι εγώ εξ αυτών ανησυχούμε για το μέλλον των παιδιών μας. Αλλά ανησυχούμε και ιδιαίτερα για τα παιδιά εκείνων που απειλούνται από πόλεμο. Δεν ανησυχούμε γιατί μπορεί να κάνουν τα παιδιά τη Συρία σε εμά. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να επενέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να ζητήσω από το Συμβούλιο να υποστηρίξει αυτή την απάντηση. Κύριε Γιούγκερ, κύριε Τίμερμαντ, η συζήτηση ω τώρα νομίζω ότι έχει καταδείξει ότι χρειαζόμαστε μια Ευρώπη η οποία θα είναι σε θέση να δράσει. Γιατί στην Ουγγαρία έχουμε κάποιε φρεχτέ εικόνε οι οποίε έχουν περάσει στην κοινωνία μα. Έχουμε ε, δει πραγματικά φρικτά γεγονότα. Αλλά να θυμάστε ότι η Ουγγαρία δεν είναι ίση με τον δίκτυο Ορμπάν. Στην ε, Ουγγαρία δεκάδε χιλιάδε πολίτε έχουν σκληρά δουλέψει για να καλωσορίσουν του πρόσφυγες. Κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι του και θα ήθελα επί τη ευκαιρία αυτή εδώ στο Κοινοβούλιο να ευχαριστήσω αυτού του πολίτε ακριβώ. Ο κύριο Όρμπαν είναι το πρόβλημα, όχι ε, τμήμα τη λύση. Η κυρία Φόρντ για ένα λεπτό, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση άνευ προηγουμένου και θα πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες σε ό,τι αφορά να βοηθήσουμε του, τη, βοήθεια στους πρόσφυγες για να φύγουν από φρικτές καταστάσεις, να τους δώσουμε ελπίδα και υποστήριξη μακροπρόθεσμα. Αλλά οι διάφορες χώρες μπορεί να βοηθήσουν με διαφορετικούς τρόπους για να σταματήσουμε να επιρρύπτουμε ευθύνε. Στον Εμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, δίνουμε πιο πολύ αρρωγή στα συριακά, στους συριακούς καταβλισμούς από ότι όλη η υπόλοιπη Ευρώπη μαζί και πολύ φοβούμαστε. Ότι θα πρέπει βασικά να κοιτάξουμε να μην ενθαρρύνουμε τη διακίνηση περαιτέρω ανθρώπων. Θα πρέπει να κοιτάξουμε ποιο είναι ο αντίκτυπος και στι γειτονικέ χώρε όταν δίνουμε άσυλο. Γιατί το να δώσουμε καθεστώς πρόσφυγα σε κάποιον δεν το δίνει αυτόματα το δικαίωμα να κινηθεί σε όλη την Ευρώπη. Αυτό θα πρέπει να είναι σαφέ γιατί η Μπορεί να υπονομεύσουμε την ε, εμπιστοσύνη του κοινού σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κινητικότητα. Να είμαστε λοιπόν ξεκάθαροι για τα δικαιώματα του κόσμου. Και ακόμα και αυτές τις δύσκολες στιγμές δεν πρέπει να υπονομεύουμε τις οικονομίες μας εκτός και αν υπάρχουν μακροπρόθεσμα Μάλλον, αν δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμα οικονομικά σχέδια υποστήριξη των χωρών μα, δεν υπάρχει μέλλον και για αυτού που χρειάζονται τη βοήθειά μα από άλλα τμήματα του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό, ο κύριο Έρνστ. Δεν είναι εδώ ο κύριος Έρνστ. Η κυρία Έρνστ. Έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι, η μετανάστευση συμβαίνει και επειδή υπάρχουν λόγοι και όσο συμβαίνει και κανείς δεν μπορεί να ορίσει ποιος ε, πρέπει και ποιος δεν πρέπει να μεταναστεύσει, δεν υπάρχουν και οι καλοί και οι κακοί πρόσφυγες όπως παρουσιάζεται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κανένα τείχος, κανένας φράχτης, καμία αστυνομική δύναμη, κανένα ρόπαλο δεν μπορεί να αποτρέψει τους ανθρώπους αυτούς. Αντί τη καταστολή η οποία εμφανίζεται συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να πούμε ένα σαφές ναι για την ενσωμάτωση των προσφύγων. Και οι πρόσφυγε θα πρέπει να πάνε και στην Ουγγαρία, στην Σλοβακία, στην Τσεχία και στην Πολωνία, σα παρακαλώ πολύ. Ανεξάρτητα από την εθνική και θρησκευτική του προέλευση απορρίπτουμε αυτή την αρχή του ασφαλούς κράτους, γιατί πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι καθόλου ασφαλείς στις χώρες της, όπως η Ρώμα στα Βαλκάνια, όπως διάφοροι στην Τουρκία. Αυτό θεωρούμε ότι είναι παράδεκτο και δεν είναι μοναδική αιτία προσφυγιάς ο πόλεμος. Θα πρέπει να τα δούμε λοιπόν αυτά και πιστεύω ότι είναι περιορισμένο αυτό. Ο κύριος Πάξας, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα ε, να παραθέσω αυτά που είπε ο κ. Σάλμποτ, ο Πρωθυπουργό τη Αυστραλία, που όταν ε, τον ρώτησαν ε, για τι προθέσει τη χώρα του για την υποδοχή παρανόμων προσφύγων από τον Παγκλαντέσσα και τη Μιανμάρ, είπε τίποτα τέτοιο δεν θα κάνουμε, γιατί αυτό θα ενθαρρύνει του υπόλοιπου να ανέβουν σε σκάφη να προσπαθήσουν να έρθουν. Αυτό θα επιδεινώσει μόνο το πρόβλημα τη παράνομη μετανάστευση. Δεν νομίζω ότι Ποιος μπορεί να ισχυριστεί πως ε, δεν εστερνίζεται ανθρώπινες αξίες ε, ο Πρωθυπουργό της Αυστραλίας. Ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας. Ε, θα έχουμε μια νέα τέτοια πολιτική η οποία θα περάσει το μήνυμα στους πρόσφυγες ότι είσαστε καλοδεχούμενοι και εδώ θα σας φροντίσουμε. Ελάτε. Ο ρυθμός των προσφύγων έχει αυξηθεί γεωμετρικά και αν δεν δράσουμε εγκαίρως και κατάλληλα, με κατάλληλο τρόπο, το μόνο που θα κάνουμε είναι να αυξήσουμε τα, τους αριθμούς περαιτέρω. Ευχαριστούμε. Για 1,5 λεπτό έχετε το... Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καλώς ορίζω την Προεδρία του Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχάς ε, για όλο το πακέτο να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κύριο Βραμόπουλο για το πακέτο το οποίο οφείλεται σε αυτόν και να τον ευχαριστήσω γιατί με τόσο σύντομο χρονικό διάστημα καταφέραμε να λάβουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο συγκεκριμένε προτάσει. Θα ήθελα κατά δεύτερον να πω ότι είναι βασικό τα πρότυπα ασύλου, τουλάχιστον τα ελάχιστα πρότυπα, να τηρούνται σε όλα τα κράτη-μέλη, προκειμένου οι πρόσφυγε, ανεξάρτητα από το που καταφθάνουν, να μπορούν να γίνονται δεκτοί και να κατανέμονται με ανθρώπινο τρόπο με μία τάξη να μπορούν να ε, γίνονται δεκτοί. Χρειαζόμαστε κατά δεύτερον ένα μηχανισμό κρίσης, γιατί χωρίς μηχανισμό κρίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αντιδράσει σωστά σε περιπτώσεις κρίσεων και σε περίπτωση ροών προσφύγων που έρχονται σε μας από πόλεμο και από ανάγκη. Κυρία Έρνστ, Υπάρχει σαφής ορισμός του πρόσφυγα και του ετούντα άσυλο. Δεν μπορούμε αυτά έτσι εθελούσια να τα μπλέξουμε με την οικονομική μετανάστευση, με τη μετανάστευση εργασίας. Θα πρέπει με σωστό νομικό τρόπο να τα ξεχωρίσουμε όλα αυτά και να δώσουμε την δυνατότητα στα κρατη ανάλογα με τις δικές τους αγορές εργασίας να αποφασίσουν ποιους θα δεχτούν. Δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε όλα τα σύνορα αντιακριτά γιατί θα ε, είχε αυτό κακά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φλέκενστάιν για ένα λεπτό. Ε, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θέλω να επαναλάβω όλα αυτά που έχουν ήδη λεχθεί. Επιθυμώ όμως ε, και εγώ να εκπέμψω ένα μήνυμα προς τις ε, τοπικές ε, κοινωνίες οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των προσφύγων υπό ιδιαίτερα αντίξωες ε, συνθήκες. Είτε πρόκειται για την ΚΟ, είτε για τη Λέσβο. Ισχύουν αυτά που σας είπα. Πόσο μάλλον για αυτούς που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρομαι στη Σερβία. Η τοπική αυτοδιοίκηση στη Σερβία κάνει για τους ε, πρόσφυγες πολλά περισσότερα από ορισμένες κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό νομίζω πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Το ίδιο λοιπόν ισχύει προφανώς ε, και για τον ε, Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, τους ε, ε, Σαμαρίτες, όπως και αν λέγονται οι διεθνείς αυτοί οι οργανισμοί και αυτούς πρέπει κάποια μέρα να τους καλέσουμε εδώ, να τους πούμε το ευχαριστώ μας γιατί ε, είμαστε πολύ πιο υπερήφανοι για αυτούς από, από ότι για κάποιους άλλους ε, πρωθυπουργού ε, της ίδιας μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόμενος ομιλητής παρακαλώ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εδώ ακούγονται πολλά ωραία λόγια, ανθρωπιά, ουμανισμός, ε, αλληλεγγύη. Ε, δυστυχώς όμως αυτά ε, πολλές φορές οδηγούν σε σύγχυση και αποδυνάμωση της Ευρώπης. Αν δεχτούμε χαοτικά παράτυπους μετανάστες οι οποίοι θα μπορούσαν να σώσουν τα παιδιά τους. Μόνοι τους τρυπάνε τις λέσβους ε, όπου μεταπνίγονται τα παιδιά. Πολλοί απειλούν ότι θα καταστραφεί το Σέγκεν. αν δεν υπάρχουν ε, ποσοστώσεις, ε, αν δεν επανεισαχθούν τα σύνορα. Μα ποιον εξυπηρετούν όλα αυτά ούτε τους ε, πρόσφυγες ούτε κανέναν άλλο απλά ε, ενισχύεται ο σκεπτικισμός εναντί της Ευρώπης. Γι' αυτό λοιπόν ας ασχοληθούμε με τα σημαντικά και να μην ε, δημαγωγούμε παρότι είμαστε πολιτικοί. Επόμενος ομιλητής και για σας παρακαλώ ισχύει το ένα λεπτό. Η κυρία δείχνει ο λαός ε, της Ευρώπης αλληλέγγυη στάση και βοηθάει τους πρόσφυγες. Αυτή είναι η Ευρώπη που θέλουμε να δούμε. Καμία σχέση δεν έχει με ε, την ε, κοινωνία των εθνικιστών και των ακροδεξιών. Αυτό το παράδειγμα πρέπει να ακολουθήσουμε. Η κατασταλτική πολιτική που μας προτείνεται δεν ταιριάζει με τις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να κάνει την επιλογή της η Ευρωπαϊκή Ένωση αν θέλει να έχει μια αλληλέγγυα ε, πολιτική για τους πρόσφυγες και για τους μετανάστες. Ε, δεν θα πρέπει να έχουμε αυξημένες ποσοστώσεις. Ε, δεν θα πρέπει να τροποποιήσουμε κατά τον τρόπο που μας υποδεικνύεται το κανονισμό του Δουβλίνου. Δεν θα πρέπει κυρίως να έχουμε ένα κατάλογο ασφαλών χωρών χωρών όπως τις χαρακτηρίζεται όπου όμως ε, αυτοί οι άνθρωποι θα διωχθούν. Δεν πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό που θέλουν οι ακροδεξιοί και οι εθνικιστές. Ε, σας ευχαριστούμε ο κύριος τώρα. Ναι, Επίτροπε, με τις προτάσεις σας απηχείτε την απίστευτη περιπλοκότητα του ζητήματος. Πρέπει να βρούμε σωστή ισορροπία ανάμεσα στην απαιτούμενη αλληλεγγύη για τους πρόσφυγες και τις άλλες χώρες, και τις ευθύνες που έχουμε και συνειδητοποιούμε ότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε και να τους σώσουμε όλους. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια ορισμένες φορές κομική συζήτηση. Κάποιοι θέλουν να έχουν καθαρή τη συνείδησή τους και άλλοι κάνουν ε, ανέφικτες προτάσεις για να έχουμε για να μηδενίσουμε το πρόβλημα της μετανάστευσης. Ε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η μαζική μετανάστευση, είναι ο άναρχος, χαοτικός, ανοργάνωτος τρόπος με τον οποίο ε, μπαίνουν στην Ευρώπη αυτές οι ροές ε, των προσφύγων. Θα πρέπει να έχουμε ένα κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών. Φυσικά πρέπει να έχουμε μια καλύτερη πολιτική επιστροφών. Φυσικά πρέπει να οργανώσουμε καλύτερα και πιο αλληλέγγυα τη διαχείριση των εξωτερικών μας συνόρων και σε διπλωματικό επίπεδο θα πρέπει να υπενθυμίσουμε σε κάποιες χώρες ότι όντως επέδειξαν γενοδορία στην υποδοχή των προσφύγων. Σκέφτομαι την Τουρκία έχει εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια πρόσφυγες ήδη υποδεχθεί όμως. Έχει κάνει και στρατηγικές επιλογές στην περίπτωση της Συρίας που είναι λανθασμένες και δυστυχώς θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο αυτό τη θέση μας. Σας ευχαριστούμε ο κύριος Βαλενσιάνου. Ένα λεπτό και για σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μεταξύ της Ελλάδας, της ε, Ιταλίας και της Ουγγαρίας τους τελευταίους μήνες έχουν ε, περάσει χιλιάδες ε, πρόσφυγες στους τελευταίους μήνες και θα πρέπει στην Ευρώπη να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό με αλληλεγγύη. Πολλές είναι η... Πολλά σωσίβια ε, λοιπόν έχουν πολύ τις τελευταίες ε, μήνες ε, και θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα λόγια της κ. Μαγκερίνη, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα λόγια πράξης τώρα, θα πρέπει να κοιτάξουμε όχι μόνο αυτές τις φρικτές εικόνες, αλλά να κάνουμε και κάτι. Θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί στην Ευρώπη. Και αυτό είναι σημαντικό. Χρειαζόμαστε λοιπόν την ειρήνη και την σταθερότητα στην Ευρώπη στο Ιράκ. Χρειαζόμαστε αποτελεσματικότητα και ειρήνη. Μόνο έτσι μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Και οι κυβερνήσεις, οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να καταδικαστούν όταν γυρνάνε και αποστρέφουν το βλέμμα σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες. Θα πρέπει να επιρρύψουμε ε, ε ποινές σε όσους δεν κινητήρουν τις αρχές μας. Ευχαριστώ. Επίτροπε, ευχαριστώ συνάδελφοι, η κυρία Γκάλα. Το ότι θέλουμε να βοηθήσουμε είναι τμήμα του DNA μας. Αυτό αφορά τη συμπόνια, αλλά θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς που πραγματικά χρειάζονται τη βοήθειά μας. Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρωτοαρχικό καθήκον είναι να προασπιστούμε τα σύνορα αυτά. Θα πρέπει να υπάρχει συνεκτικότητα και αυτό βλέπω να λείπει από τις δράσεις ως τώρα. Μια συνεκτικότητα και εφαρμογή των κανόνων που υπάρχουν. Αν δεν τα καταφέρουμε αυτά, θα καταρρεύσει το Σέγγεν. Οι κανόνε του Σέγγεν για τα εξωτερικά σύνορα, οι όροι υπό του οποίου επιτρέπεται κανεί να μπει στο Σέγγεν, ισχύουν αυτοί οι κανόνε. Ήθελα να ξέρω. τι γίνεται και με του κανόνε για την ε, επιστροφή στον πρώτο κράτος μέλος ε, που καταφτάνει ο, ο Αν αυτά ισχύουν, πώς ε, μπορούμε να κατηγορούμε την Ουγγαρία που εφαρμόζει απλά τους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί. Προσπαθεί απλά να προσπιστεί τα εξωτερικά σύνορα η Ουγγαρία. Οι πιο πολλοί που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να θυμάστε. Και διακόπτει ο Πρόεδρος. για ένα λεπτό. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ακούσαμε ε, σήμερα το πρωί από τον πρόεδρο κύριο Γιούνκερ που έκανε αναφορά σε αυτούς τους καλούς ανθρώπους στο σταθμό του Μονάχου ε, και τους καλούς ανθρώπους στα ελληνικά νησιά. Κύριε Επίτροπε, και εσείς ε, Έλληνας είστε, βλέπουμε καλούς ανθρώπους ε, και στη δική μου τη χώρα και αλλού, αλλά εγώ ρωτάω κάτι το πολύ απλό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει και η δική μου απάντηση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τελικά το άθροισμα των κρατών μελών ε, που βεβαίως πρέπει να το πω και αυτό θα συναντηθούν επιγόντω τη Δευτέρα. Εκεί λοιπόν να δείξουν ότι τα προγράμματα που παρουσιάστε σήμερα ε, είναι σοβαρά, ότι θα εφαρμοστούν. Το Κοινοβούλιο έχει κάνει τη δουλειά του να υπάρχει ταχύτατη ανακατανομή. Εμείς κάναμε τα μαθήματά μας. Αυτά όμως ε, που θα γίνουν τη Δευτέρα είναι σημαντικά. Τι θα γίνει τη Δευτέρα, θα ρίχνει ο ένας τον μπαλάκι στον άλλον ή μήπω θα δούμε μια πραγματική αντίδραση στην ε, κρίση αυτή, τη μεγαλύτερη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το άθροισμα των πολιτών γι' αυτό στις 14 Σεπτεμβρίου είτε θα πετύχουν όλοι μαζί είτε θα κατακριμνιστούν. Ε, κοντριτσο παρακαλώ ένα λεπτό και για σας. Κύριε Πρόεδρε, ε, το θέμα δεν είναι ότι έχουμε να κάνουμε μόνο με το πρόβλημα της μετανάστευσης στο νότο της Ευρώπης και κλείνουμε τα μάτια σε αυτά που συμβαίνουν στο ανατολικό κομμάτι της Ευρώπης. Όχι, ξέρουμε ότι στο, ε, στα σύνορα μεταξύ Ντόμπρατς και Ρωσίας ε, και εκεί πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι αγωνίζονται και αγωνιούν οι άνθρωποι για τη ζωή τους και η ζωή δική τους κινδυνεύει και όχι μόνο των ε, Σύριων η Πολωνία Εφαρμόζει λοιπόν μια συνειδητή πολιτική όπου ε, κάθε χρόνο δεχόμαστε πάνω από ένα εκατομμύριο Ουκρανούς και τους δίνουμε και θεώρηση, βίζα. Ήδη φέτος έχουν φτάσει και έχουν ζητήσει βίζα πάνω από 500.000 Ουκρανοί στην πατρίδα μας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή η πολωνική ελληνική κυβέρνηση να ανοίξει και για πρόσφυγες από τον Νότο, αλλά κάτω από προθέσεις που θα μας επιτρέπουν να τι αντιμετωπίσουμε με αξιοπρέπεια. Η κυρία Μουσολίνη. Κύριε Γιούγκε, είναι σημαντικό να τροποποιηθεί η συνθήκη του Δουβλίνου για να αντιμετωπιστεί το ανθρωπιστικό δράμα. Αυτό ισχύει για την Ιταλία και για τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Αυτό το λίγο και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Τέλεια. Πολύ σύντομη. Και έτσι λοιπόν ε, μπορέσαμε να έχουμε κάποιο χρόνο πριν από την ψηφοφορία και έτσι μπορούμε και να περάσουμε στη διαδικασία Catch the Eye τουλάχιστον μία παρέμβαση αναπολιτική ομάδα. Κυρία, μάλλον Κέλλη, για ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριος Κέλλη. Ε, νομίζω ότι η αλληλεγγύη και όλες αυτές οι αξίες είναι αξίες ε, που αναφέρθηκαν από τον ε, πρόεδρο Γιούνκερ σήμερα, αλλά αντικατατουρίζονται και από όλη την Ευρώπη. Και σίγουρα η Ιρλανδία συμμερίζεται αυτές τις αξίες και ε, είναι έτοιμη να υποδεχτεί πιο πολλούς πρόσφυγες. Δύο ερωτήσει. Είπατε για την υποδοχή από οικογένειες. Αυτό μπορεί να ε, ενσωματωθεί στην ευρωπαϊκή πολιτική και ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κεφάλαια. Κατά δεύτερον, ο πρόεδρος Τάσκ δικαίως καταδίκασε τους διακινητές ως δολοφόνους. Αναρωτιέμαι μήπως μπορεί να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση τους, να κατάσχουμε τα πλοία τους, γιατί αυτοί είναι οι πραγματικοί θήτες και θα αυτούς θα πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σλάνγια, η κυρία Σλάνγια, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, τον Απρίλιο ψηφίσαμε επί ενό ε, ψηφίσματο που ήδη ζήταγε δεσμευτικέ ποσοστώσει για να καταμερίζονται καλύτερα ευθύνε ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Το 2014, 6 από τα 28 κράτη-μέλη μόνα του διαχειρίστηκαν το μεγαλύτερο ποσοστό των αιτήσεων ασύλου στην Ευρώπη. Ίσως αυτό λοιπόν να είναι η αλληλεγγύη, ε, γιατί αυτό αναφέρεται και στα σχετικά άρθρα τη συνθήκη. Πιστεύω λοιπόν ότι η συμπεριφορά του ε, Συμβουλίου είναι καταδικαστέα ε, η δική μου πρόσκληση είναι να κάνουμε βήματα προς τα μπρος, αυτά που αποφασίσαμε ήδη τον Απρίλιο, ε, αυτά που είπε η Κομισιόν να εφαρμοστούν, να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός ε, για την τήρηση των ποσοστώσεων. Έχουμε ευθύνες ως Ευρωπαίοι και γι' αυτό πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτές. Υπάρχει περιφερειακή αστάθεια και υπάρχουν και ανισότητες. Σας ευχαριστώ πολύ. Τζαμπάνσκι ε, για ένα λεπτό και εσείς Πρόεδρε, θα πρέπει καταρχήν να υπάρχει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στους πρόσφυγες και τους παράτυπους μετανάστες όσοι έρχονται στην Ήπειρό μας ε, τον αντιμετωπίζουμε ως ε, πρόσφυγα ε, θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε προστασία σε πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους που έρχονται από την Αφρική και τη Μέση Ένα πολύ σημαντικό είναι να μιλήσουμε για τα αίτια της μετανάστευσης τα αίτια έχουν σχέση με τον πόλεμο που εξακολουθεί να μένεται στη Συρία και στο Ιράκ υπάρχουν συγκρούσεις και σε άλλες χώρες στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή. Έτσι λοιπόν ε, ε, αν συνεχιστούν τα πολιτικά παιχνίδια σε αυτές τις χώρες οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να ε, φεύγουν. Όσοι λοιπόν είναι κατά του ISIS θα πρέπει να στηριχθούν, να χρηματοδοτηθούν και να υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Επόμενος ομιλητής, Μπιλμπάο, ε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε αυτή την κρίση των προσφύγων χρειαζόμαστε συγκεκριμένα γεγονότα και πράξεις. Εμείς ε, στη χώρα των Βάσκων προσπαθούμε να επιδείξουμε αλληλεγγύη. Στις 14 Σεπτεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή πολιτική που να βασίζεται στην αλληλεγγύη και την υπευθυνότητα. Ως εκ τούτου οφείλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στην αποδοχή των μεταναστών, να τα οργανώσουμε όλα αυτά ε, σε σαφείς ε, ατραπούς που να οδηγούν προς την Ευρώπη και να καταπολεμήσουμε και τη μαφία που μπλέκεται και αυτή με τους μετανάστες. Σωστή λοιπόν αποτελεσματική πολιτική στις χώρες προέλευσης και επίσης ε, σωστή πολιτική κατανομής. Ε, με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα αίτια που οδήγησαν στο να αντιμετωπίζουμε τις μεγαλύτερες ροές προσφύγων από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εμείς ως Βάσκοι προσπαθήσαμε αυτής εξ αρχής να βοηθήσουμε. Επόμενος ομιλητής επίσης για ένα λεπτό. Κυρία Σακοράφα. Κυρία Σακοράφα παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η σημερινή μακροσκελή και θαραλέα, θα έλεγα, εισήγηση του Προέδρου Γιούγκερ, που έστω και περιγραφικά αναφέρεται στι αιτίε και στι ευθύνε Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί την πιο επίσημη ομολογία αποτυχία τόσο τη εξωτερική όσο και τη προσφυγική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δυστυχώ γίνεται υπό το βάρο χιλιάδων νεκρών και απάνθρωπων συνθηκών διαβίωση για του πρόσφυγε και την πίεση που αντιμετωπίζουν πλέον οι χώρε τη κεντρική ευρώπη. Κύριοι συνάδελφοι, έστω και την τελευταία στιγμή, α αντιμετωπίσουμε ολοκληρωμένα το τραγικό ανθρωποκτόνο ζήτημα με παράλληλε και αποτελεσματικέ δράσει σε όλα τα επίπεδα. Αναγνωρίζοντα πρώτα απ' όλα τι ευθύνε μα και μη επιτρέποντα ξανά να υπάρξει κανένα άλλο πρόσφυγα πνιγμένο ή νεκρό. Κανένα πρόσφυγα σε άθλιε συνθήκε διαβίωση, με αλληλέγγυα αξιοπρεπή αντιμετώπιση τη ανθρώπινη υπόσταση, διασφαλίζοντα ότι η βοήθεια προ του πρόσφυγε θα αποτελέσει ευθύνη του συνόλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με άμεση εξασφάλιση νόμιμη πρόσβαση και ασφαλών διαδρομών με θέσπιση μηχανισμού μετεγκατάσταση με μόνιμο και υποχρεωτικό χαρακτήρα με την κατάργηση του κριτηρίου τη χώρα τη πρώτη εισόδου με ουσιαστικέ και αποτελεσματικέ πρωτοβουλίε για την εμπόλεμε περιοχέ και Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε στον επόμενο μιλητή ε, που θα μιλήσει για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν ήμουν σε κίνδυνο θα ήθελα και εγώ να φύγω. Αυτή είναι μια σαφής αρχή την οποία και γνωρίζουμε, όμως η διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι το άσυλο είναι ε, το να ε, μπορεί κανείς ε, χορηγείται όταν υπάρχει πολιτική δίωξη και υπάρχει και σαφής ορισμός των οικονομικών μεταναστών. Οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι προτάσεις της εγκαταλείπουν αυτές τις αρχές των ΗΕ. Προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει διεθνές δίκαιο και θέλει να καταργήσει τη συμφωνία του Δουβλίνου. Η μεσαία τάξη και οι εύποροι που έχουν την ικανότητα και τη δυνατότητα δυνατότητα να ε, ξεφύγουν από προβλήματα αγνοούν τους φτωχούς, αυτούς που δεν έχουν φωνή, αυτούς ε, που είναι αναγκασμένοι να ζουν διάσπαρτοι στην ε, Ευρώπη και να υποφέρουν από τις συνέπειες. Δεν μπορεί κανείς να έχει κατά νου μόνο τους μεν και να ξεχνάει τους δε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος Μορβάη, παρακαλώ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω απολύτως με την κυρία Γκάλ. Θα ήθελα να ρωτήσω, μάλλον θα ήθελα να ζητήσω η σημερινή συζήτηση και η ψηφοφορία να μην οδηγηθούν ε, στην κατάσταση όπου δεν θα έχουμε μια ικανοποιητική απάντηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε δεσμευτικά πρότυπα. Ε, τα συμμορφώνεται ναι ή όχι η Ουγγαρία με αυτά. 15 εκατομμύρια Ούγγροι περιμένουν μια συγκεκριμένη απάντηση από εσά και νομίζω ότι την ίδια απάντηση περιμένουν ε, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες πώς θα υπερασπιστούμε τα σύνορά μας. Δώστε μας μια ξεκάθαρη απάντηση. Η κυρία Μέρκελ ουσιαστικά έχει απευθύνει πρόσκληση σε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι την ε, αντιλαμβάνονται. Θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα να έρθουν στην Γερμανία. Και ε, τους εμποδίζουν κάποια αστυνομικά μέτρα δεν θέλουν να πάνε στα κέντρα μεταναστών και προσφύγων, ε, δεν θέλουν να συμμορφωθούν ε, με την νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί τι πρέπει να κάνουμε, τι περιμένετε από εμά. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος, κλείνει εδώ η συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ που τηρήσατε το χρόνο. Σε κάποιους έκοψα αγενώς ε, το λόγο, αλλά τι να κάνω, δεν γινόταν αλλιώς. Τώρα λοιπόν θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Αβραμόπουλο. Παρακαλώ κύριε Αβραμόπουλε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους σας για αυτά που είπατε και για την γενικότερη υποστήριξή σας προς την προσέγγιση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πραγματικά ελπίζω οι προτάσεις μας να υιοθετηθούν χωρίς καθυστέρηση γιατί τώρα πια χρειαζόμαστε ταχύτατα αποφάσεις. Προσβλέπω ιδιαίτερα στη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις επικείμενες συζητήσεις για το μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης. Και επίσης ε, και τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου ε, στον κατάλογο των ασφαλών κρατών. Εκεί το Κοινοβούλιο θα είναι συνομοθέτης. Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εφαρμόσουμε τις αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί και να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα εφαρμόζουν τους κοινούς ε, κανόνες. Και βεβαίως ε, θέλουμε να υπολογίζουμε στην στη στήριξη του Κοινοβουλίου σε αυτές μας τις ε, προσπάθειες. Γιατί ξέρετε αυτή η μετανάστευση θα διαρκέσει. Αυτό είναι γεγονός. Το πακέτο το οποίο υιοθέτησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μόνο μόνο ένα βήμα για την καλύτερη διαχείριση της ε, μετανάστευσης. Έχουμε επίσης ακόμα πολλή δουλειά για την ε, αφομοίωση των μεταναστών. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για να υπάρχει πολιτική συνοχή. Μια επιτυχής ε, πολιτική για τη μετανάστευση είναι καθοριστική σημασίας η συνεργασία με τις τρίτες χώρες και το άνοιγμα νόμιμων οδών και αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Αυτό βεβαίως συμβαδίζει με τον πόλεμο που έχουμε κηρύξει απέναντι στους ε, αντίστακτους διακινητές. Τα κρατημέλη έχουν συμφωνήσει επί ενός ε, προγράμματος μετεγκατάστασης ε, Ποτέ παλιά δεν είχε συμβεί αυτό να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε 22 περίπου χιλιάδες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να βασιστούμε λοιπόν σε αυτή την επιτυχία και να αναλάβουμε στο μέλλον και άλλες πρωτοβουλίες για να υπάρχουν νόμιμες δυνατότητες να έρθει κανείς στην Ευρώπη. Και τέλος είναι καθοριστική σημασία να προστατεύονται τα σύνορά μας. Εμείς λοιπόν θα αναλάβουμε πρωτοβουλία για να ενισχύσουμε την καλύτερη διαχείριση των σύνορων μας για να υπάρξουν φιλόδοξες λύσεις. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας. Κατέγραψα τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας και με χαρά διαπίστωσα ότι όλοι μας έχουμε μια κοινή φιλοδοξία να συνεργαστούμε, το κάναμε κατά το παρελθόν, να το κάνουμε και κατά το μέλλον, να υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση και τέλος σε κοινέ λύσεις. Πραγματικά προσβλέπω στη συνεργασία, στη συνέχιση ε, της ε, συνεργασίας μας, αυτής που είχαμε ήδη κατά τους τελευταίους μήνες. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Ο Επίτροπο μίλησε εκ μέρου ε, τη Επιτροπή, Τώρα το λόγο στο Συμβούλιο ο Υπουργό Κύριο Σμίτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν πολύ πλούσια η συζήτηση και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Λουξεμβουριανή η Λουξεμβουργιανή Προεδρία, όπως είπε και ο Επίτροπος, θα συνεχίσει αυτό το διάλογο και τη συνεργασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρακαλώ ησυχία συνάδελφοι. Γιατί ολοκληρώνονται μια πολύ σημαντική συζήτηση. Το λόγο λοιπόν έχει το Συμβούλιο και θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους να καθίσουν, να ακούν προσωπικά, να κάνουν ησυχία. Ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη. Έλεγα λοιπόν ότι θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία και ο διάλογος με το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο Γι' αυτό το πολυσύνθετο ζήτημα στη δύσκολη στιγμή στην οποία βρισκόμαστε. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σημειωθεί τάχιστα πρόοδος, νομίζω το ακούσατε από όλου τους ενδιαφερομένους και θα εργαστούμε επί τη βάση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το επόμενο Συμβούλιο που θα λάβει χώρα την Δευτέρα φέρει μια μεγάλη ευθύνη από αυτή τη πλευρά και πραγματικά ελπίζω ότι η πληθώρα των μηνυμάτων που ακούσαμε στις παρεμβάσεις σας ε, θα ληφθούν δεόντως υπόψη ε, κατά τη διάρκεια των εργασιών του επομένου Συμβουλίου. Υπάρχει μία συνένεση βάσει της οποίας ε, πρέπει να συσπηρωθούμε και να είμαστε σαφείς ως προς τις προτεραιότητες μας αλλά και τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να επιτύχουμε στους στόχους μας για να μπορέσουμε να επιτύχουμε σε αυτό το εγχείρημά μας. Ταυτόχρονα θα πρέπει να συμφωνήσουμε για τα νέα εργαλεία που είναι προσαρμοσμένα στη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Χρειαζόμαστε μια σφαιρική προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε την κρίση και επαναλαμβάνω αυτά που σας είπα στην αρχική μου παρέμβαση. Δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε, ε, πρέπει να αποφύγουμε κάθε παρελκυστική συμπεριφορά διότι δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Σμιτ. Ευχαριστώ βεβαίω ε, εξ ονόματο όλων των συναδέλφων, το Συμβούλιο και την Επιτροπή που ήρθαν σήμερα εδώ σε αυτή την τόσο σημαντική συζήτηση. Και θέλω να σα ανακοινώσω ότι έλαβα 7 προτάσει ψηφίσματο μετά την ολοκλήρωση τη συζήτηση για τη μετανάστευση. Η συζήτηση έκλεισε και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στι 12. Και τώρα λοιπόν για σήμερα, για την ε, ψηφορία. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο κύριο Βίλαντ. Οι αρμόδιε ελληνικέ αρχέ ε, μα ζήτησαν την άρση σας.